ενίσχυση της τρομοκρατικής απειλής. Θα παρακαλέσω τον ε, Υπουργό κύριο Μπέρτ Κούντερς να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Επί τη ευκαιρία αυτή, δέκα εβδομάδες μετά τις ε, επιθέσεις στις τρομοκρατικές στο Παρίσι, θέλω να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναζήσουμε στην Ευρώπη τέτοιες τρομερές επιθέσεις. Θα ήθελα να μπορώ να το πω, αλλά δεν είμαι πεπισμένος. Αντίθετα, βάσει των πρόσφατων ε, γεγονότων και πληροφοριών βλέπουμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί κομμάτι της Ευρώπης και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην ε, πιο κοντινή μας γειτονιά, αν λάβουμε υπόψη μας ε, την Κωνσταντινούπολη, το Χασαντά, το Πακιστάν, ο Αγαντούγκου κλπ. Ως Προεδρία λοιπόν εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις και να προστατεύσει τους πολίτες. Ο αντιτρομοκρατικός αγώνας θα αποτελέσει το κέντρο τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε με τους αρμόδιους υπουργούς του Άμστερνταμ. Επίσης η Προεδρία δίνει μεγάλη σημασία στο κράτος δικαίου και προκειμένου να έχουμε μια καλή ισορροπία στην, στον αγώνα μας αυτό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, υπάρχουν εμπόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε για την τρομοκρατία. Και το ξέρουμε αυτό και θα είναι στην ατζέντα μα. Ένα άλλο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών όσον αφορά τα πυροβόλα, όπλα και τα εκρηκτικά. Η εφαρμογή των μέτρων που συμφωνούνται είναι στοιχείο κλειδί για να πετύχει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-2020. Επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων έκαναν δήλωση για την αντιτοκρομοκρατία το Φεβρουάριο του 2015 μετά από τις επιθέσεις στο Σαρλί Εμπτό. Και αυτή ακριβώ η δήλωση αποτελεί και το πλαίσιο που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σε εφαρμογή και να υλοποιήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί και η Ευρωπαϊκή Προεδρία για να πετύχουμε. Πολλά έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και υπάρχουν σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συντονιστή της δηλαδή, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συνεργασία μεταξύ μας είναι στοιχείο κλειδί και αυτό το έχει εντοπίσει το Συμβούλιο. Έχει επιτευχθεί πρόοδος μέχρι τώρα. Υπάρχει συμφωνία για την οδηγία για το ευρωπαϊκό PNR, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε εν δυνάμει τρομοκράτες. 1η Ιανουαρίου η Europol ξεκίνησε με το κέντρο της κατά της τρομοκρατίας. Είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν οι διάφορες χώρες. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στην έρευνα όσον αφορά του ξένους μαχητές και τη χρηματοδότηση των ε, αυτών. Θέλουμε να βοηθήσουμε επίσης τους εμπειρογνώμονε στο ΣΥΤΙ προκειμένου να προχωρήσουμε τη δικιά του ομάδα εμπειρογνωμόνων για την έρευνα τέτοιων δράσεων. Τέτοιε έρευνε γίνονται σε πολλές χώρε μέλη. Επίσης, ελέγχουμε και την συνεισφορά όλων των χωρών με δεδομένα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκτός τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί υπάρχουν επαφές και ανταλλαγή πληροφοριών με τους ομολόγους μας των υπηρεσιών πληροφοριών σε τρίτες χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει και πρόταση όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών για εγκληματίες. Επιπλέον αρχίσαμε να συζητάμε και την πρόταση για να τροποποιηθεί η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Σεπτέμβριο η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο οδηγία. ώστε να λάβουμε υπόψη μας και το ψήφισμα 2178 του ΟΗΕ. Οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία αυτή έχουν ήδη προχωρήσει και πιστεύω ότι τον Ιούνιο θα μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα οριστικό. Τώρα πέρα από τις πληροφορίες όσον αφορά την συμμόρφωση προς τον νόμο, η επιτυχία μας είναι το βασικό. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, ξέροντας πόσες χιλιάδες ε, πολίτες Ευρωπαίοι έχουν φύγει για να πάνε να πολεμήσουν στη Συρία. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, διακρίσεις, ευκαιρίες πρέπει να υπάρχουν για όλους. Πρέπει να υπάρχει ανοχή, να υπάρξει ε, θρησκευτικός διάλογος, διαθρησκευτικός διάλογος και εμείς προσβλέπουμε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόληψη όμως δεν φτάνει από μόνη της. Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλά εκπαιδευμένοι μαχητές οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν απειλή. Οι βέλτιστες πρακτικές είναι αυτό που πρέπει να προωθήσουμε και έχει γίνει πολλή δουλειά μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να μάθουμε ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ και να μιλήσουμε με πυρογνώμονε από όλε χώρε και να μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία μα αυτή και σε τρίτε χώρε, στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Αφρική και την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο είναι μία από τις κύριες πηγές ενημέρωσης για τους ανθρώπους αυτούς, τους φανατικούς. Στα πλαίσια λοιπόν του κέντρου αντιτρομοκρατίας της Europol γίνεται δουλειά και προς αυτή την κατεύθυνση για να αντιμετωπιστούν οι τρομοκρατικές απειλές. Από 3 Σεπτεμβρίου του 2015 υπάρχει και το δίκτυο, το φόρουμ αυτό της Ευρώπης με περιεχόμενο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται σε συνεργασία με τους παρόχους. Η συζήτηση τώρα για ένα πρόγραμμα δράσης κατά του λαθρεμπορίου όπλων είναι και αυτό κάτι που προχωράει. Η Προεδρία συμφωνεί με την προσέγγιση. Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στο πακέτο των, ε, της φύλαξης των συνόρων. Οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθούν. Είναι πρώτη προτεραιότητά μας η ασφάλεια. Δεν πρέπει βέβαια με τίποτα να μπερδεύουμε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την απειλή, αλλά μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι μετανάστες προσπαθούν να φύγουν από τον πόλεμο, από μέρη όπου διώκονται και να προστατεύσουν τους αυτούς τους και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δέσμευση που έχουμε ήδη αναλάβει και με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Αφρική. Όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και έχει αποδειχτεί αυτό και με το δικό σας το ψήφισμα, το περσινό, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τόσο αποφάσισε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς η Επιτροπή σας λείπει. Προσβλέπω σε καρποφόρα συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κούντες. Τώρα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έχει το λόγο. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ. Thank you, Mr. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. κύριε Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε το 2015 ήταν ε, <clears throat> κομβική χρονιά για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ένιωσε την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία στέρισε τη ζωή 150 αθώων πολιτών. Πολλές ζωές χάθηκαν λοιπόν <clears throat> και πάρα πολλές ζωές φοβήθηκαν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλή. Η τρομοκρατική απειλή είναι παρούσα. Είμαστε αποφασισμένοι να απαντήσουμε με ανθεκτικότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τις αξίες, τις δικές μας αξίες ανοχής, δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την εργασία της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Μερίσια Διάταξη για την Ασφάλεια <clears throat> ξέρετε ότι έχει τεθεί προς συζήτηση ήδη από τον προηγούμενο Απρίλιο έχουμε ξεκινήσει την ταχύτατη προσπάθεια εφαρμογής και για το Ευρωπαϊκό PNR σαν παράδειγμα. Έχουμε κάνει την πρόταση για μια οδηγία για την τρομοκρατία. Το Νοέμβριο υπήρξε το πακέτο για τα μικρά όπλα. Ε, τέθηκε επίσης το θέμα του προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των όπλων και τα κέντρα αριστείας για την καταπολέμηση της ρισοσπαστικοποίησης, όπως επίσης και η εκκίνηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ στο διαδίκτυο. Και την εβδομάδα αυτή η πρόταση για την ανταλλαγή των ποινικών μητρών. Όλα αυτά είναι απτά μέτρα θα έλεγα, τα οποία έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την ασφάλειά μας ε, διαμεθοριακά και θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Το 2016 θα είναι η χρονιά όπου θα κυνηγήσουμε το χρήμα των τρομοκρατών. Απαιτείται να στερήσουμε τους τρομοκράτες από τους οικονομικούς τους πόρους. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα καταθέσουμε επίσημα τις προτάσεις μας με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πακέτο για, για τα σύνορα του προηγούμενου Δεκεμβρίου είναι καθοριστικό στοιχείο του παζλ γιατί θα επιτρέψει τον συστηματικό έλεγχο ασφαλείας όλων αυτών οι οποίοι εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> και ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι απαιτείται να βελτιώσουμε τη διαχείριση των εξωτερικών μας σύνορων για να βελτιώσουμε την εσωτερική ασφάλεια και να διασώσουμε το Σέγγεν. Θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρος για μια ακόμη φορά για ένα σχετικό θέμα. Οι πρόσφυγες οι οποίοι περνούν τα σύνορά μας διότι χρειάζονται διεθνή προστασία και δικαιούνται διεθνή προστασία δεν είναι τρομοκράτες. Πρέπει να το επιβεβαιώσω, να πω ότι ποτέ δεν θα εξισώσουμε τους πρόσφυγες με τους τρομοκράτες. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αφήσουμε να κυριαρχήσει ο φόβος. Τώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά όπως γνωρίζετε κρίσιμο θέμα. Όπως γνωρίζετε επίσης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ημερήσιας διάταξής μας στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά μέσα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Schengen, η, τα δεδομένα και οι τράπεζες βάσης ε, της ε, Interpol θα πρέπει, της Europol συγγνώμη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπιστεύονται περισσότερο το ένα το άλλο. Θα πρέπει να μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους αλλά και με τη Europol. Οι δυνάμεις επιβολής τάξης στα διάφορα κράτη-μέλη, ακόμα και οι εξοδικευμένες υπηρεσίες, συνεργάζονται και έχουν όλες τον ίδιο στόχο, την ασφάλεια δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι συλλογικά είμαστε ασφαλέστεροι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνδυάσουμε ε, την απάντησή μας και την ανταπόκρισή μας στις απειλές. Δεν έχουμε να κάνουμε με εσωτερικό ανταγωνισμό, Απλά αν συνεργαστούμε ε, θα είμαστε αποτελεσματικότεροι. Ήδη υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα, αλλά χρειάζεται να αυξηθεί και όχι να μειωθεί. Την επόμενη εβδομάδα επίσημα θα ξεκινήσουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας στην Europol. <clears throat> Λειτουργεί ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Το κέντρο αυτό νομίζω ότι θα είναι το κέντρο, η πλατφόρμα του συνδυασμού των ενεργειών μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εφόσον το χρησιμοποιήσουμε σωστά και εφόσον τα κράτη-μέλη πράγματι μοιραστούν τις πληροφορίες. Το κέντρο αυτό θα πετύχει την αποστολή του, στην αποστολή του, εφόσον το βοηθήσουμε. Πρέπει λοιπόν να το στηρίξουμε, πρέπει να δούμε ότι η βοήθεια της Europol στους Γάλλους και τους Βέλγους ανακριτές μετά τις επισκέψεις στο Παρίσι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου, η διασταύρωση των στοιχείων, η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και η παροχή αναλυτικών και λειτουργικών τρόπων βοήθειας και αρρωγής προς τις εθνικές υπηρεσίες. Είναι οι στόχοι της υπηρεσίας αυτής. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου μετά από τις επιθέσεις στο περιοδικό Σαρλί Εμπτό υπογραμμίσαμε ότι η απάντησή μας δεν θα χαρακτηριστεί από τον φόβο και το μίσος ή τα βιαστικά συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες είναι τμήμα μιας συναλλικής ανταπόκρισης. Στα πλαίσια αυτής της συλλογική προσπάθειας νομίζω ότι έχει υπάρξει πρόοδος. Τα τελευταία γεγονότα όμως μας υπενθύμησαν ότι απαιτείται να κάνουμε πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι τώρα έχει πλέον έλθει η στιγμή της δράσης και της ενίσχυσης των μορφών συνεργασίας μας. Ας είναι το 2016 ένας κονδικός χρόνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αποτροπή τέτοιου είδου καταστροφών στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Βόζεμπεργκ να λάβει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το περιοδικό Ντάμπια με τον τίτλο Just Terror γράφει επιλέξει Let Paris be a lesson for those nations. Το Παρίσι να γίνει μάθημα για, τα, για εκείνους που πρέπει να καταλάβουν. Και δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες των τρομοκρατών που χτύπησαν στο Παρίσι τις προάλλες, σημαίνει ότι θέλουν να διαφημίσουν μια πολιτική της τρομοκρατίας. Η πολιτική της τρομοκρατίας όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περάσει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπνέεται από τις αρχές και τους κανόνες της πολιτικής της δημοκρατίας σήμερα σύμφωνα με τις έρευνες της europol περίπου έξι χιλιάδες πέντε χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες είναι τρομοκράτες. αυτό θα το επιτρέψουμε να συνεχίζεται; πώς μπορούμε να το ελέγξουμε; τι έχει κάνει η ευρωπαϊκή ένωση και το συμβούλιο; έχουμε κάνει βήματα πολύ σημαντικά και η απάντηση στους τρομοκράτες είναι ότι ο φόβος δεν μπορεί να επικρατήσει. πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο όμως να ελεγχθεί; υπάρχουν οι δομημένες ομάδες υπάρχουν τα δίκτυα των τρομοκρατών υπάρχουν στόχοι και οι στόχοι αφορούν σε ανθρώπινες ζωές στην περιθωριοποίηση της ευρώπης στο κλείσιμο των συνόρων. είναι πολύ ορθή η πολιτική την οποία ακολουθούμε και δεν μπορούμε να συγχέουμε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση το ένα φαινόμενο με το άλλο ανεξάρτητα αν με την ανεξέλεγκτη ροή των ε, μεταναστών πολλές φορές παρισφραίουν και τρομοκράτες. δεν υπάρχει περίπτωση όμως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή ένωση η ευρωπαϊκή αντίληψη να συνδυάζει αυτά τα δύο φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να το προσέξουμε πολύ σοβαρά είναι πώς θα ελέγξουμε το φαινόμενο. Θα το ελέγξουμε μέσα από το διαδίκτυο, θα το ελέγξουμε μέσα από την συνεργασία των κρατών μελών, θα το ελέγξουμε μέσα από τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διότι η τρομοκρατία έχει πρόσωπο, το πιο απεχθές πρόσωπο, στο οποίο η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γιούρεκ την δέχεστε παρακαλώ το μικρόφωνο του ομιλητή δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο του ομιλητή ωραία σας ευχαριστώ πολύ και στα δικά σας λόγια και τα λόγια του Επιτρόπου Αβραμόπουλου ακούω πολλά αληθινά και πολύτιμα σχόλια. Δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε την ε, ε, μετανάστευση, την προσφυγιά με την τρομοκρατία ή να θεωρήσουμε ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Δεν πιστεύετε όμως ότι το να έρθουν εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη αποτελεί βάση για την ανάπτυξη της τρομοκρατίας γιατί είναι ένα ε, ευρωπαϊκό φαινόμενο και εξαγόμενο. Κύριε συνάδελφε, εφόσον δεν συνδυάζουμε τα δύο φαινόμενα θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ευρώπης και γι' αυτό δουλεύει η ευρωπαϊκή ένωση ούτως ώστε τέτοια φαινόμενα να αποτραπούν. ο δρόμος της αποτροπής των ανθρώπων να έρχονται στην ευρωπαϊκή ένωση δεν μας χαρακτηρίζει. η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να ελέγχει τα εξωτερικά της σύνορα αλλά η διακίνηση των πολιτών των εμπορευμάτων μέσω της σέγγεν και των ιδεών είναι μέσα μέσα στις αρχές που διαπνέουν ακριβώς την ένωση τη δική μας. σας ευχαριστώ. Η κυρία Σίπλε λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες δεν κατευθύνονται κατά συγκεκριμένων ανθρώπων. Στόχο έχουν να διαχύσουν τον φόβο και ως εκ τούτου να διαταράξουν τη δημοκρατία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Χρειάζονται σαφείς τοποθετήσεις κατά της τρομοκρατίας και άμυνα των κοινωνιών μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι η τρομοκρατία δεν είναι αυτή τη στιγμή εθνικό φαινόμενο και ως εκ τούτου θα πρέπει τα ευρωπαϊκά μέσα για την αξιοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών να αξιοποιηθούν προληπτικά. Η τρομοκρατική προπαγάνδα μέσα από το ίντερνετ πρέπει να ε, ανοιχνεύεται, πρέπει να γίνονται έρευνες εις βάρος των τρομοκρατικών δηλώσεων μέσα από το ε, διαδίκτυο και άλλων. Πρέπει να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση και τα σχετικά δίκτυα με συστήματα ε, συμβουλών και προληπτικά και καλούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν αντίστοιχα την επάνδρωση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ανάλογα με τις, δυνα... ανάγκες για να μην υπάρχουν κενά. Χρειάζεται και ψηφιακά και αναλογικά να ενισχυθούν οι δικαστικές ε, διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ορισμοί για την ποινική περιγραφή των αδικημάτων της τρομοκρατίας. Το ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Και πάντα πρέπει δικονομικά να έχουμε ασφαλή αποδεικτικά στοιχεία. Πρόληψη λοιπόν, ανείχνευση, δίωξη και καταδίκη. Με τα βήματα αυτά μόνο μπορούμε να διαφυλάσσουμε και την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και έτσι αποτελεσματικά να, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Ευχαριστώ, και ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα ξεκάθαρα να πω ότι η τρομοκρατική απειλή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκέ μας χώρε. Έχουν δυστυχώς υποτιμηθεί η κίνδυνη από την ε, ριζοσπαστικοποίηση και βέβαια έχουν αποτύχει οι πολυπολιτισμικές ε, κοινωνίες ε, και λόγω των ακραίων πολιτικών χωρών όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και άλλες που είναι χορηγοί τέτοιων οργανώσεων. Ο Πρόεδρος, σας επισημαίνω ότι μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Ναι, μάλιστα, λέει ο μιλητής. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να ε, δίνουμε ε, επένους και οικονομικούς όπως συνέβη με την Τουρκία σε αυτούς που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις αυστηρές. Ιδάλλως η τρομοκρατία θα μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Λιέζεκ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η τρομοκρατία έχει σαρώσει ζωές, αξίες, τρόπο διαβίωσης. Ευρύτατο είναι το φάσμα της απειλάς και γι' αυτό απαιτείται ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή συνεργασία και ανταπόκριση, συνεργασία βέβαια με τους εταίρους μας όλο τον κόσμο. Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση είναι ένα συμμετροϊκό ε, πόλεμο θα πρέπει να εστιάζεται στα εξή θέματα. Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και ρίζα της τρομοκρατίας, ρίζες και αίτια της τρομοκρατίας. Πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά λοιπόν την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, πρέπει να ε, ελέγξουμε καλύτερα τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες που με τόση ευκολία κάνουν ένα κατά του Παρισιού ε, όπως οι προπληρωμένες κάρτες ε, πρέπει να κοιτάξουμε τα δίκτυα της διακίνησης και του λαθρεμπορίου πρέπει να κοιτάξουμε μέτρα σε κάθε επίπεδο τοπικό μέχρι και πανευρωπαϊκό και βεβαίως τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά χωρίς να είναι υπερβολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία μεταξύ ε, αστυνομίας και άλλων ε, υπηρεσιών δίωξης και επιβολής της τάξης θα πρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά. Δεν επιτρέπεται να παραλάβουμε τα ασφάλματα του παρελθόντος. Βέβαια πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ύψιστη, η, ε, ο ύψιστος ο βαθμός της επαγρύπνησης. Δεν πρέπει κανείς να μπαίνει ή να βγαίνει από την Ευρώπη, από τους συνοριοφυλακές και τις ακτοφυλακές. Είναι αυτός άλλωστε και ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και το λαθρεμπόλιο όπλων και η πρόσβαση των τρομοκρατών στα όπλα. Ωστόσο, αυτό είναι μακράς πνοής. Ε, υπάρχει και μακράς πνοής καθήκων. Αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ευρώπη και έφτασαν να γίνουν μαχητές ε, ε, για την τρομοκρατία, προδίδοντας τις ίδιες τους τις πατρίδες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό θα πρέπει να γίνει με μέτρα και προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ζήμπερα ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στρατηγική της ε, αντιμετώπισης ε, της τρομοκρατίας προβλέπει τον περιορισμό των προσωπικών δικαιωμάτων και η απάντηση γενικά είναι μιλιταριστικού τύπου και ενισχύει τη λογική αντιπαράθεσης μίσους και πολέμου. Τα μέτρα αυτά τα οποία έχετε προτείνει υπονομεύουν τις ατομικές ελευθερίες και είναι ένα τμήμα γενικά της στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων και της παρεμβατικότητας που οδηγεί σε ξενοφοβία, ρατσισμό και τρομοκρατία στην Ευρώπη. Φρικτά εγκλήματα σαν και αυτά τα οποία συνέβησαν στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές του κόσμου απαιτούν μια ειρηνική απάντηση, ε, το απαιτούν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου ε, και ενίσχυση των ειρηνευτικών προσπαθειών. Έτσι μόνο θα αντιπαρατεθούμε στην τρομοκρατία. Ο κύριος ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. άκουσα ότι η Προεδρία υπογραμμίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε σε λύσεις απέναντι στο πρόβλημα ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν, γιατί τα κράτη-μέλη ήταν υπεύθυνα για την ανυπαρξία κοινών μέτρων ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις ειδικές περί υπηρεσίες και ενίσχυση της Europol και άλλων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύστημα δεν δουλεύει ακόμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα σχετικά με υπόπτους, με κινδύνους και απειλές. Στην ουσία συλλέγουμε εκατομμύρια δεδομένων για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και παρεμποδίζουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι, και για καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Εξακολουθούμε να ζούμε σε δημοκρατίες που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τους κανόνες της δημοκρατίας και αυτό το υπενθύμησε και το δικαστήριο του Στρασβούργου για μια συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση από την Ουγγαρία που έλεγε ότι για να διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και όχι απλά να συλλέγονται στοιχεία χωρίς κανένα λόγο. Ο κύριος Βούλφ. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο βασικός κανόνας για τη λειτουργία μιας κυβέρνησης είναι η προστασία του λαού της. Η προστασία των λαών της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο κατανοούμε και είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όμως της τρομοκρατίας πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους συνομιλούμε και αν συμμερίζονται τις αξίες μας. Και εκεί η ανάλυση σας αποτυγχάνει. Για να κατανοήσετε το πρόβλημα πρέπει να κατανοήσετε τον αντίπαλο. Και το πρώτο επίπεδο είναι ότι και στη δική σας ρητορική και στη ρητορική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπατε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών ξεφεύγουν από την τρομοκρατία. Όχι βέβαια. Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών είναι οικονομικοί μετανάστες. Αυτοί που ζητούν άσυλο είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν. Πρέπει να κάνετε τη διάκριση λοιπόν. Το δεύτερο τμήμα του προβλήματος είναι ότι τα ανοιχτά σύνορα τα οποία δημιουργήσατε και δεν θέλετε να αφισβητήσετε δεν σας επιτρέπουν να γνωρίζετε ποιος έρχεται και ποιος είναι και πού πάει. Και αυτό γεννά την τρομοκρατία, την εσωτερική τρομοκρατία την οποία οι γυναίκες στη Σουηδία, στο Βερολίνο, στην Κολομία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης αντιμετώπισαν και θα αντιμετωπίζουν. Υπάρχει μπλε κάρτα για σας. Δέχεστε από τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Τη μετάφραση περιμένετε. Ωραία. Τώρα, καταλάβατε. Εντάξει τώρα. Μπορείτε να θέσετε την ερώτησή σας στα αγγλικά μήπως. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, είπατε πολλά και συμφωνώ μαζί σας, αλλά Συμφωνείτε και εσείς μαζί μου για το ότι η τρομοκρατία είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο, γιατί τρομοκρατία έχουμε και μέσα στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε Βόρεια Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι δικό μας ευρωπαϊκό πρόβλημα. Πρόκειται για, τον για την ευρωπαϊκή τρομοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην μιλάμε λοιπόν μόνο για τρομοκρατία που μας έρχεται απ' έξω στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα παγκόσμιο φαινόμενο η τρομοκρατία και νομίζω ότι πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Όλες τις μορφές τρομοκρατίας πρέπει να καταπολεμήσουμε. Συμφωνείτε μαζί μου. Είναι εξαιρετικά τα αγγλικά σας. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να καταλάβω και να μιλήσω τη δικιά σας γλώσσα τόσο καλά. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Όντως, είναι διεθνές πρόβλημα η τρομοκρατία πονάει και πλήττει οικογένειε ολόκληρο τον κόσμο. Και ναι, έχουμε προβλήματα και εδώ με του Ευρωπαίου στη δικιά μα βάση στην Ευρώπη. Όμω αυτό που συζητάμε σήμερα είναι εκείνο του ISIS. Είναι μια ιδεολογία η οποία τα βάζει τους ανθρώπους να παλεύουν μεταξύ τους άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες επίση Γι' αυτό χρειάζεται μια συνολική λύση και είναι ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Μάγερ, τώρα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να αναφερθώ και εγώ στην τρομοκρατική απειλή και δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήσει ότι η Ευρώπη είναι στόχος των τρομοκρατών. Είχαμε στο Παρίσι, αλλά όχι μόνο και στις Βρυξέλλες, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο. Δεν ξέρουμε όμως γιατί έγιναν αυτά, γιατί δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε τίποτα από όλα αυτά και να τα αποφύγουμε εμπνέονται από το Κοράνι οι άνθρωποι αυτοί που προχωρούν σε τέτοιε τρομοκρατικέ επιθέσει. Γι' αυτό θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα όλου αυτού που μπαίνουν στην Ευρώπη. Και παρά τη μεγάλη απειλή που έχουμε εδώ στην Ευρώπη, παρόλα αυτά η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι μια ουτοπία. Νομίζει ότι θα μπορέσει να αποφύγει την τρομοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Το Ισλάμ είναι αυτό που φταίει, που κυριαρχεί στα μυαλά των ανθρώπων αυτών. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε αυτήν την πολιτική ανοιχτών ε, συνόρων που έχει σαν αποτέλεσμα η Ευρώπη να γίνεται βάση για αυτούς τους τρομοκράτες. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, να αποφύγουμε δηλαδή αυτή την ε, παρέμβαση, αυτή την εισβολή που έχουμε απ' έξω στις χώρες μας με τόσες χιλιάδες που πέρασαν από την Ελλάδα για παράδειγμα, που ήταν και τσιχαντιστές μερικοί από αυτούς. Αυτή όλη είναι απειλή και είναι απειλή και για τις γυναίκες. Συνεπώς πρέπει να ξαναδούμε το Σέγγεν. Τα ανοιχτά σύνορα τελικά δεν έχουν βοηθήσει. Αντίθετα, μπορούμε να περιμένουμε και άλλες μαζικές επιθέσεις αν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. Ενώ πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική ασφάλειας για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Η μόνη λύση είναι να κλείσουν τα εθνικά σύνορα. Και όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως ε, ετούντες άσυλο τελικά θα οδηγήσουν στον Ισλαμισμό της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φουντούλης τώρα για ένα λεπτό. Ξαφνικά η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία. Τόσο το κίνημά μας η Χρυσή Αυγή όσο και άλλα εθνικιστικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το ότι πρόκειται να συμβεί. Μας κατηγορείτε για Ισλαμοφοβικούς. Πείτε το αυτό στους γονείς των παιδιών που πήγαν στον Πατακλά να διασκεδάσουν και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους δεν θα υποκύψουμε λέτε στην τρομοκρατία όταν πρωτεύουσε ευρωπαϊκών χωρών έχουν το στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπίσουν την απειλή. έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του ευρωπαίου πολίτη. οι πολιτικές σας των ανοιχτών συνόρων της κατάρρευσης των αξιών και του πρωτοφανούς ρατσισμού εις βάρος των γηγενών δεν μπορούσαν παρά να προσφέρουν γόνιμο έδαφος στο σπόρο του ισλαμικού φονταμεταλισμού όσο και να προσπαθείτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να το αποκρύψετε η τρομοκρατία στην ευρώπη έχει ισλαμική ταυτότητα. η οργανωμένη επίθεση στην κολονία την πρώτη του έτους εναντίον γυναικών είναι τρομοκρατικό χτύπημα. έστειλαν το μήνυμα είμαστε εδώ και θα αποσιωπητικά τις γυναίκες τις κόρες και τις αδερφές σας και εσείς προτείνετε στις γυναίκες να μην ντύνονται προκλητικά να μην φορούν αρώματα. τα περισσότερα τζαμιά που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην ευρώπη δεν είναι παρά φυτώρια τρομοκρατών. ποια είναι η λύση; εγκαταλείψτε τις ιδεολογικές σας αγκυλώσεις θωρακίστε την ήπειρό μας από τα εκατομμύρια που κάθε χρόνο παράνομα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και για τις προσπάθειες που από κοινού κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε με προβλεπτικότητα και αξιοπρέπεια το μεγάλο δράμα των τρομοκρατικών μορφών βίας στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τα νέα τον τελευταίο καιρό δεν είναι ικανοποιητικά, δυστυχώς Νομίζω ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πούμε ότι η δράση την οποία αναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γύρω από το θέμα του PNR και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και μια προσπάθεια για την κοινή άμυνα, οδεύουν προς την καλή κατεύθυνση, τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν. Η αναπόφευκτη αδυναμία μας είναι σε πάρα πολλούς τομείς δυστυχώς και επηρεάζουν αρνητικά και την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού της μετανάστευσης επίσης. Αρνούμεθα εμείς να συνδέσουμε την τρομοκρατία με τη μετανάστευση. Φυσικά είναι λάθος να συνδέουμε τα δύο φαινόμενα συστηματικά. Είναι επίσης λάθος να αγνοούμε ότι τα δύο φαινόμενα έχουν κοινά αίτια οι Ισλαμικές περιοχές παράγουν τρομοκρατικά φαινόμενα σαν αυτά τα οποία με δραματικό τρόπο έφυξαν την Ήπειρό μας και το μέτωπο στο οποίο δυστυχώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Κοράνι σαν όπλο και θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ε, θα μεταφέρουμε την δημοκρατία εκεί που δεν υπάρχει. Η αποσία της δημοκρατίας, η απουσία του πολιτισμού την οποία εμείς έχουμε σαν κληρονομιά του χριστιανικού παρελθόντος μας γεννούν την τρομοκρατία. Φαγιών. Κύριε Πρόεδρε, όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερες τρομοκρατικές δραστηριότητες εκδηλώνονται στον κόσμο, στην Πουρκίνα Φάσο, το Πακιστάν, παντού. Και θα κοιτάμε κάποτε τη χρονιά 2015 με μεγάλη θλίψη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ε, είναι οι αποκλεισμένοι των κοινωνιών που οθούνται προς την, ε, προς την ακρότητα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τους πρόσφυγες από τους τρομοκράτες. Οι περισσότεροι πρόσφυγες φεύγουν από τις χώρες τους λόγω των τρομοκρατών. Και αν δεν ενισχύσουμε τα μέτρα ασφάλειας και την ασφάλεια δεν θα τα καταφέρουμε. Χρειάζονται όμως και κοινωνικά μέτρα. Χρειάζεται να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να καταπολεμηθεί η ρίζα του κακού. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ξεκάθαρη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Ανταλλαγή πληροφοριών, ναι, βεβαίω είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι ότου συμβεί αυτό, κανένα μέτρο δεν θα είναι αποτελεσματικό και γι' αυτό θα πρέπει να οικοδομήσουμε το την εμπιστοσύνη, να ανταλλάσσετε πληροφορία και στοιχεία, να διαγιγνώσκεται η πορεία των όπλων και του χρήματος και με εξέπληξε το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε μέσα στη νέα νομοθεσία PNR την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει πολλές τραγωδίες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστική μουσουλμανική προπαγάνδα, την αξιοποίηση των μέσων μαζική ενημέρωση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε του γονεί να λύσουμε την, απαραίτη, την απαιτούμενη ε, την απέτηση μάλλον για ε, άδεια από τους γονείς όταν τα παιδιά τους ταξιδεύουν ε, στο εξωτερικό και όλα αυτά. Αλλά μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος, ε, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ρουζαντόφσκι εκεί πάνω ψηλά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε και κυρία συνάδελφε. Αν δεν απατώμε, σοσιαλιστές ήταν εκείνοι που αρνήθηκαν την επιτάχυνση των εργασιών της οδηγίας PNR. Τώρα ξέρουμε ότι έχει καταθέσει μια νέα πρόταση μιας αντιτρομοκρατικής οδηγίας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς εσάς απευθύνω το ερώτημα, μια και είσαστε σοσιαλίστρια, έχετε σοσιαλιστική ομάδα, θα υποστηρίξει η ομάδα σας τη νέα πρόταση της Επιτροπής ή θα έχουμε την ίδια παρεμπόδιση που είδαμε στο PNR. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτησή σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Απαιτείται βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε και να ε, παραβιάσουμε κάθε έννοια προσωπικού και ιδιωτικού βίου. Χρειάζεται η ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει η πρόταση και τι θα ε, ανταλλάσσεται ως πληροφορία. κυρία Φανστόρχ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, μιλούμε για την τρομοκρατία, την απειλή, το Παρίσι, την κολονία. 338 καταγγελίες, 30 ύποπτοι, περισσότεροι από αυτούς ε, πρόσφυγες, 11 από αυτούς είχαν μόλις μπει τον Δεκέμβριο στη Γερμανία. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε μόνο για κρίση μεταναστών. Ένας από τους δράστες είχε, του Παρισιού ήταν και αυτός είχε περάσει μέσα από τα δίκτυα των, ε, της προσφυγιάς. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι είναι τρομοκράτες, αλλά οι τρομοκράτες που βρίσκονται μεταξύ αυτών, που συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών, καταχρώνται των δομών μας και είναι υπερβολική πια η αριθμή τους. Και η διαπερατότητα των συνόρων μας τους διευκολύνει. Ο κύριο Σέχοφερ στη Γερμανία μιλάει πολύ. Η Τσέντεου γράφει πολλές επιστολές. Η καγκελάριός μας θα μείνει στην ιστορία ως αυτή που διέλυσε την Ευρώπη, ακόμη και αν παρατηθεί πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Παγαθαουρτουντούα Ρουίχτ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν για τα αρμοδιότητες που πρέπει να αναλάβει ο καθένας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και πολύ ωραία, πολύ καλά πάει αυτό και σας ευχαριστούμε που υπάρχει συνοχή. Όμως υπάρχουν και αδυναμίες. Από αυτά που είπατε εγώ δύο αδυναμίες βλέπω κυρίως. Πρώτον, ότι όταν πρόκειται για μια συνολική απειλή δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται. Δεν συνεργάζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα, με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτή είναι μια μεγάλη αδυναμία. Γιατί όσοι συνδεόμαστε, οι υπηρεσίες μας δηλαδή συνδέονται μεταξύ τους και έχουν ανταλλαγή, είναι πολύ καλό. Το δεύτερο είναι η πρόληψη. Και αυτή είναι αδυναμία, ότι δεν υπάρχει έγκαιρα πρόληψη σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ποιε είναι οι καλέ πρακτικέ και ποιε όχι. Εσεί τι θα κάνετε, θα κάνετε μια έρευνα επειδή κάπου υπάρχουν ευέλτιστε πρακτικέ. Πιο συστηματικοί πρέπει να είμαστε. Σε τοπικό επίπεδο, από εκεί να αρχίσουμε. Έτσι θα αποφύγουμε τα προβλήματα. Και πρέπει να δουλέψουμε και περισσότερο εκεί που υπάρχει η μεγάλη αδυναμία, που είναι ακριβώ αυτό που σα είπα, η πρόληψη, η έγκαιρη πρόληψη. Δέχεστε μπλε κάρτα, παρακαλώ. Κύριε Μισόνη. Ο κύριο Σόνι έχει μπλε κάρτα. Είναι δεξιά σα. Δεξιά σα. Α, έτσι. Εκεί. Τον βλέπετε. Παρακαλώ. Κύριε Σόνι. Σόνι. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία συνάδελφοι, αναφερθήκατε σε δύο προκλήσεις Έχω μια τρίτη να σας ε, προτείνω. Δεν ανησυχείτε για το ότι ορισμένες κυβερνήσεις μπορεί να αντιδρούν υπερβολικά. Θα αναφέρω την Ουγγρική κυβέρνηση η οποία θέλει να εισαγάγει καθεστώς ε, κρίσεως. Και πώς ε, αξιολογείται αυτή την αντίδραση των κυβερνήσεων. Είναι λογική, είναι αναλογική. Απάντηση. Πολύ χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Ένας από τους κινδύνους, από τους πειρασμούς, είναι οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν το φανατισμό, τους ε, τρομοκράτες. Πάνε πέρα από τον νόμο, βγαίνουν από τον νόμο. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να τιμωρούμε τους υπεύθυνους, αλλά σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, γιατί αλλιώς θα έχουμε χάσει τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Το κράτος δικαίου πρέπει να τηρείται. Ο νόμος να υπάρχει όχι ατιμορρησία, αλλά βάσει του νόμου. Αλλιώς είναι μπούμεραγκ. Ευχαριστούμε κύριε Γκονζάλης τώρα ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν χρειάζεται μαθήματα για τις ελευθερίες μας και τα δικαιώματά μας. Είμαστε μπροστά σε μια πρόκληση που για την οποία για να την αντιμετωπίσουμε οφείλουμε να προχωρήσουμε βάσει της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο μέσα στα σύνορά μας όσο και εκτός. Πρέπει να κοπεί η χρηματοδότηση, η βοήθεια λογιστική προς το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους δημοκράτες στην Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο. Πρέπει να εξουδετερωθούν τα δίκτυα εκείνα τα οποία φέρουν τρομοκράτε. και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με την ταξί των υπηρεσιών πληροφοριών. Πρέπει να προστατεύσουμε όμως χρόνο τους πρόσφυγες, οι οποίοι θέλουν ακριβώς να φύγουν από την τρομοκρατία. Πρέπει ο κόσμος να νιώθει μέρος μιας κοινωνίας και να βοηθήσουμε κοινωνικά και οικονομικά τους πιο αδύναμους. Πολλοί τρομοκράτες έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο καταπολεμείται μόνο με πολιτικές βοήθειας και εκπαίδευσης. Η κυρία Σαρτζαντίνη τώρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ακούω τον Επίτροπο να κάνει κάποιες προτάσεις για το τι θα κάνουν για να σταματήσει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, προτείνουν κάποια πράγματα. Όμως πρέπει να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Γιατί όταν έχετε στις 11 ε, Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, στην Νέα Υόρκη, ε, την τρομοκρατία ή στην ε, Βοστόνη, την τρομοκρατική επίθεση ή στο Παρίσι. Όλα αυτά δεν κοστίζουν πολλά χρήματα. Άρα δεν είναι το θέμα της χρηματοδότησης από τον ΤΑΣ. Στη Συρία τώρα, στη Μέση Ανατολή, από ό,τι φαίνεται, πληρώνονται οι άνθρωποι για εκεί οι μαχητές από το ίδιο το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Οπότε χρειάζεται να βρούμε τα ίχνη αυτών των ε, δικτύων δεν είναι θέμα πολλών χρημάτων. Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα για τρομοκρατία, έστω και με τα λίγα χρήματα αυτά που τους χρειάζονται. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν ακριβώς, πώς ακριβώς θα πετύχετε αυτά που λέτε. χρησιμοποιούν και ένα παλαιού τύπου φεουδαλικό κατάλοιπο τρόπο μεταφοράς των χρημάτων από το ένα μέρος στο άλλο. Φεράρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αύξηση της τρομοκρατικής απειλής δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην απίσχναση των δημοκρατικών δικαιωμάτων ε, και των δημοκρατικών αξιών. Η ευθύνη πολέμησης του φαινομένου αφορά βέβαια κυρίως τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει έτσι ώστε να υπάρξει ένας αποτελεσματικός διάλογος ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών κάθε κράτους αλλιώς θα οδηγηθούμε στην επανεισαγωγή των ε, ελέγχων στα σύνορα, τα εσωτερικά πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να μην συνεχίσουμε να συλλέγουμε τυφλά όλο και περισσότερα δεδομένα, αλλά να είμαστε επιλεκτικοί, να εντοπίσουμε τους τρόπους τροφοδοσίας των τρομοκρατικών οργανώσεων, δεν είναι κάτι το ανέφικτο, απαιτείται η πολιτική βούληση. Μπονάνο 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εκπρόσωπο της Ολλανδικής κυβέρνησης. Εκφράζω την, την οργή μου γιατί είμαστε 751 εδώ και τώρα βλέπουμε ότι οι υπάλληλοι είναι πιο πολλοί από τους βουλευτές. Τι είδου Ευρώπη είναι αυτή που θέλει να λύσει ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα. Μου τη δίνει λέει ο, ο μιλητής, μου τη σπάει λέει ο μιλητής. Ντρέπομαι για τον ευρωπαϊκό λαό, ε, σαν ακροκόδιλοι κλαίμε για αυτά τα οποία συνέβησαν στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στη Νέα Υόρκη και η απάντησή μας ποια είναι. Α, οι Ισλαμικές, οι Ισλαμιστές φταίνε, η τρομοκρατία φταίει. Τώρα αυτά είναι ντροπή πράγματα. Αυτή η Ευρώπη δεν υπάρχει. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να βοηθήσει τους Ευρωπαίους. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ζόμπι. Είμαστε όλοι ζόμπι. Οι εχθροί έχουν τα πάντα και θα επιτεθούν και ο λαός της Ευρώπης θα υποστεί τις συνέπειες. Και εμείς τι λέμε, ευχαριστούμε στο Ισλάμ. Δίνουμε κάτι δισεκατομμύρια στην Τουρκία, ενώ γνωρίζουμε ότι το 90% των Τούρκων είναι Ισλαμιστές. Λοιπόν, το πρόβλημα μου δεν είναι οι Ισλαμιστές, αλλά είμαστε Ευρωπαίοι, ανήκουμε στη Δύση. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος διακόπτοντας τον κύριο Μπονάνο. Έχετε δύο μπλε κάρτες. Θα τις δεχτείτε. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς είναι ο πρώτος που θα σας θέσει την ερώτηση. Θα το πω στα Ιταλικά για να με καταλάβετε πιο εύκολα. Μήπως ε, τελικά περισσεύει η υποκρισία. Όταν εσείς έρχεστε στην Ολομέλεια εδώ ε, μόλις τώρα μπήκατε στην αίθουσα και αμέσως μετά από αυτό που είπατε θα φύγετε. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ από το πρωί ως το βράδυ. Και όπως είπε ο Σαλβίνη, ε, ε, είναι κρίμα να μην είναι εδώ ο πρόεδρός σας μάλλον, είναι κρίμα να μην είναι παρόντες οι βουλευτές και μετά αμέσως φεύγει. Λοιπόν αυτό δεν είναι παρά υποκριτικό. Κοιτάξτε, σε αυτούς που χειροκροτούν θα τους πω να κοιτάξουν τα δεδομένα μου. Στους 751 είμαι στην 17η θέση για την παρουσία μου στην Ολομέλεια και τη συμμετοχή μου στις ψηφοφορίες. Αυτά μην μου τα λέτε εμένα. Εγώ έρχομαι εδώ, δουλεύω, είμαι στη 17η θέση και είμαι και δήμαρχος. Εσείς λες ότι είσαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρεις εγώ τι κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια ερώτηση τώρα από την κυρία Ευχαριστώ. Ναι, εσεί δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει τρομοκράτε. Εγώ ναι. 13 χρόνια, επειδή είχε δολοφονηθεί ο αδερφό μου, ζούσα με αστυνομική προστασία. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε θεάματα, άλλες και είμαστε στο θέατρο. Πρέπει να υπάρχει πνεύμα συνεργασία. Εσεί αναφερθήκατε σε μια Ευρώπη των ζόμπι. Εγώ δεν είμαι ζόμπι. Εγώ έρχομαι εδώ να δουλέψω και να προσφέρω ό,τι μπορώ. Όχι φανατισμό. Ξέρω πώ φανατίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Έχω γνωρίσει τρομοκράτε διαφόρων ειδών. Δεν χρειάζεται να μας βρίζετε και να μας προσβάλλετε επειδή είμαστε εδώ που συζητάμε και δεν υπάρχουν ίσως και πολλοί οι οποίοι λένε νοησίες, αλλά υπάρχουν και υπόλοιποι οι οποίοι μιλάνε σοβαρά και προσπαθούν να δουλέψουν και να βοηθήσουν. Και σας το λέω εντελώς καλοπροαίρετα. Ευχαριστώ. Ε, Εγώ δεν τα έχω βάλει μαζί σας γιατί είστε παρούσα και δεν ανήκετε σε αυτούς τους οποίους ασκώ κριτικής, πόσο μάλλον. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ε, κυβερνούν την Ευρώπη δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά, δεν θα ασχολούνται με τα θέματα των Ισλαμιστών στην κολονία και τους βιασμούς. Θα φανούν αδιάφοροι και όλοι αυτοί οι οποίοι χειροκροτούν εδώ σαν μικροί πίθηκοι, θα καταλάβουν ότι στην ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν τη μουσική που τους επιβάλλουν οι υπόλοιποι. Κύριος Παπαδάκης, ένα λεπτό. Πλέον υπάρχει μεγάλη πείρα στους λαούς. Από τους Μουτζαχεντίν, τον Μπιν Λάντεν, την Αλκάιντα ως το Ισλαμικό κράτος ανατράφηκαν όλοι τους από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μοναρχίες του κόλπου για τα συμφέροντά τους αποτελούν διαχρονικά για τα συμφέροντά τους ε, το βολικό πρόσχημα για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης. σπέρνετε τις αραβικές ανοίξεις που εξελίχθησαν σε βαρχημονιά για τους λαούς και θερίζεται με ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αποκαλούμενες αντιτρομοκρατικές εκστρατείες με πολυπλόκαμους μηχανισμούς καταστολής και φακελώματος σκόπιμα η ευρωπαϊκή ένωση επιχειρεί να τσουβαλιάσει τον ριζοσπαστισμό των λαών όπως και τους πρόσφυγες με την τρομοκρατία και να ενισχύσει το νομικό της οπλοστάσιο απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα για να βάλει στο γύψο τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες για να ενοχοποιήσει τον αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που υπερασπίζεται απέναντι στη βάρβαρη εργατική επίθεση που προωθούν η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσεις τους είναι προδιαγεγραμμένο ότι οι λαοί θα ξεσηκωθούν. σαν το αποφασίσουν θα δείξουν τη δύναμη τους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χολμάιρ. Δυόμιση λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα επί του κανονισμού να πω κάτι πρώτα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο, όταν εκφράζονται από βουλευτές ε, προσβολές εις βάρος ηγετών κρατών και κυβερνήσεων να τους ε, διακόπτεται, γιατί δεν είναι αυτός τρόπος να ε, συνομιλούμε. Επί της ουσίας τώρα. Η τρομοκρατία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές, κυρίες και κύριοι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και εγώ 20 χρόνια είχα συνοδεία σωματοφυλάκων και απειλές είχαν εκφραστεί αντίον της οικογένειάς μου. Ξέρω πολύ καλά πώς αισθάνεται κανείς που βρίσκεται υπό τη μόνιμη απειλή. Αλλά εδώ η τρομοκρατία έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Στρέφεται κατά του κάθε ενός εκείνου ο οποίος δεν ακολουθεί την παράφρονα, ε, τις παράφρονες επιλογές της, ε, του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους. Αυτούς που πάνε να χορέψουν, αυτούς που πάνε να ακούσουν μουσική, να κάτσουν να φάνε σε ένα εστιατόριο, απλώς να λιαστούν. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κενά εκείνα τα σχετικά με την καλώς νοωμένη προστασία των δεδομένων στην νομοθεσία ώστε να γίνεται σωστά η ανταλλαγή των πληροφοριών. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και τα δεδομένα Eurodac, Eurodac να μπαίνουν μέσα στα μητρώα των δραστών και να μην μπορεί κανένας τρομοκράτης να περνάει κρυμμένος ως πρόσφυγας σύνορα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους εμποδίζουμε να μπαίνουν σε αεροπλάνα ή σε ροές προσφυγικές. Και βεβαίως η αμοιβαία αναγνώριση στις δικαστικές και άλλες διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτατα. Η ε, κατάδικοι θα πρέπει να καταγράφονται σε μητρό πανευρωπαϊκά ώστε να μην μπορεί κανείς να ε, ξεφεύγει από τους ελέγχους αστυνομίας. Πρέπει να ενισχυθούν οι αστυνομικές δομές αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται για να μας προστατέψουν από τους τρομοκράτες. Δεν μπορούμε μόνο να τους επισημαίνουμε διαρκώς τα λάθη τους. Πρέπει να τους ενισχύουμε και ηθικά και σημειώνω ότι σε αυτό είναι πολύ εύκολο να ε, κατακρίνει κανείς, είναι πολύ πιο εύκολο να κατακρίνει από το να αναλάβει να κάνει την ίδια δουλειά ο ίδιος. Στο PNR, προστασία δεδομένων και σχετικές οδηγίες, Πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να στερέψουν οι πηγές της χρηματοδότησης. Μία από τις αιτίες ή από τις πηγές που οδηγούν στην εκδήλωση τρομοκρατικών επιθέσεων. Και έτσι μπορούμε νομίζω να έχουμε χτίσει κάτι αποτελεσματικό κατά της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Τζαμπάσκι. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφο. Τι θέση έχετε για τις ε, πληροφορίες που έχουν διαθέσει η Γερμανία αστυνομική και διαδόθηκαν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι τους δόθηκαν οδηγίες να αποκρύψουν την προέλευση των ε, δραστών των επιθέσεων της κολονίας την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τι θέση έχετε γι' αυτό. Πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει η διερεύνηση ενός εγκλήματος και όχι να καταδικαστεί μία εθνικότητα. Εάν η εθνικότητα έχει συμμετοχή ως για να σιουργώσει αιτία σε ένα έγκλημα, τότε ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι η εθνικότητα ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε συγκεκριμένα εγκλήματα. Εγώ θέλω να γίνεται διερεύνηση των εγκλημάτων και όχι να κοιτάω πού είναι η, πιανού είναι η υπηκότητα, η εθνικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν περιοχές που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε non-go, απαράβατα, ε, μέρη όπως το Μόλεμπεκ, όπως άλλες περιοχές απο, απομονωμένες, οι οποίες δεν μπαίνουν οι δυνάμεις της τάξεως. Ο Πρόεδρος. Δεύτερη μπλε κάρτα. Από τον κύριο Κράσινο Τέψικη. Τη δέχεστε. Ναι, θα ρωτήσω λοιπόν τα εξή. Πώς αξιολογείται το γεγονός ότι τα γεγονότα της κολονίας δεν δημοσιοποιήθηκαν τις πρώτες ημέρες, δεν βγήκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έγινε ο δημόσιος διάλογος. Είπε ο κύριος Τζεμπάνσκι ότι δόθησαν εντολές στην αστυνομία να συγκρατήσει τις πληροφορίες αυτές. Αλλά εν γέννη ούτε η κοινωνία της Γερμανίας ούτε εκείνη η γνώμη ευρύτερα στην Ευρώπη είχε ενημερωθεί. Όλα αυτά που συστούμε εδώ πώς μπορούν να βοηθήσουν την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος της τρομοκρατίας δηλαδή. Ναι, ακούστηκαν επικρίσεις για το ότι ένας ε, κρατικός σταθμός μόνο δύο μέρες μετά ενημέρωσε το κοινό για τα γεγονότα. Όλοι οι άλλοι όμως είχαν αμέσως ενημερώσει. Και επίσης πιστεύω ότι εάν εγκαίρως είχαμε μπορέσει να μπούμε σε περιοχές ε, άβατες, αυτές τις non-go areas, ε, όπως το Μόναχο συμβαίνει, θα είχαμε αποτρέψει αυτά τα αδικήματα, θα είχαμε εμποδίσει την οργάνωση των ε, δραστών και δεν θα είχαμε προβλήματα. Γιατί ακριβώς εκεί έγινε το πρόβλημα, στα no-go areas. Ευχαριστώ, Νίτερ Μίλλερ. Πρόεδρε. Τα γεγονότα του Παρισιού έσπηραν το φόβο αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε την ψυχραιμία μας, την ελευθερία, τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Πρέπει να μην ανοίξουμε πεδίο διάδοσης ε, και διάξης ακόμη περισσότερο του φόβου, όπως προσπαθούν να πράξουν τα ε, λαϊκιστικά κόμματα. Δεν υπάρχει καμία τρομοκρατική απειλή που να δικαιολογεί την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών. Πρέπει να αναλάβουμε βήματα για να πατάξουμε οποιονδήποτε στρέφεται κατά της δημοκρατίας μας. Δηλαδή να εμποδίσουμε αυτό ακριβώς που θέλουν και οι τρομοκράτες όπως και οι λαϊκιστές να περιστήλουν τα δικαιώματά μας και τις ελευθερίες μας. Είμαστε της ε, άποψης ότι η δημοκρατία, τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να τύχουν προστασίας. Κανένα κέρδος δεν έχουμε από τις μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών. Χρειάζεται απλώς καλύτερη συνεργασία, χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών. Και ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε, να μην αφήσουμε περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση της, των μεταναστών της δεύτερης και τρίτης γενιάς, δηλαδή να προσφέρουμε κατάρτιση, εκπαίδευση, ενσωμάτωση, πραγματικές προοπτικές στην Ευρώπη, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η ενσωμάτωση στις κοινωνίες δεν ισοδυναμεί με αφομοίωση, αλλά ότι ταυτόχρονα δεν υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με την ένταξη την κοινωνική και την κοινωνική ενσωμάτωση. You have a blue card from Mr. Jurek. You accept... Μπλε κάρτα από τον κύριο Γιούρεκ. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ρωτήσω, ο λαϊκισμός, ο εξτρεμισμός, αυτή η γλώσσα δεν οδηγάει στον αποκλεισμό. Είναι γλώσσα μίσους. οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν δημοκρατικά εκλεγμένοι. Εσείς πιστεύετε ότι όταν συνεχίσουμε να μιλάμε με αυτή την γλώσσα θα καταλήξουμε σε κοινωνικό διάλογο, για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση που είχε ποτέ η Ευρώπη. Μαζί πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Στην μπλε κάρτα σας ανακοινώνω ότι δεν θα δέχομαι δεύτερη μπλε κάρτα στον ίδιο ομιλητή. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η σημερινή συζήτηση νομίζω δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι μιλούν για τρομοκρατία, απειλές και πρόληψη. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν τη συζήτηση για να εκδηλώσουν απόψεις κατά του Ισλάμ, κατά της μετανάστευσης, κατά των προσφύγων. Πιστεύω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο δεν χρειάζονται τέτοιες τοποθετήσεις. Πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα και για, τα αντικειμενικά πραγματικά γεγονότα. Ο κύριος Νίκολσον. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ότι το 2015 μας παρέπεμψε στα πολύ σοβαρά προβλήματα της τρομοκρατίας ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος με τα σύνορά μας, για τα σύνορά μας, ιδιαίτερα τα σύνορα Σέγγεν, και πουθενά στην Ευρώπη δεν είναι ασφαλές, ε, ασφαλής ο τόπος μετά από αυτά που συνέβησαν. Εγώ φυσικά προέρχομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία, ξέρουμε την τρομοκρατία, επιβίωσα μια τρομοκρατικής ε, απόπειρα εις βάρος μου. Δεν είμαι ζόμπι όμως, να πω στον προλαλήσαντα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δακτυλοδεικτούμε. Ε, τα θύματα της τρομοκρατίας δυστυχώς τα ξεχνάμε συστηματικά μετά από αυτό το οποίο συμβαίνει περνάμε στην επόμενη φρικτή ενέργεια, στο επόμενο έγκλημα και αγνοούμε τις συνέπειες της προηγούμενης. Απαιτείται λοιπόν στην Ευρώπη να υπάρξει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών και απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας και διασυνοριακά ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής. Για ένα λεπτό, η κυρία Ευχαριστώ. Είναι συνολική παγκόσμια τρομοκρατική απειλή τόσο μέσα όσο και έξω από την Ευρώπη. Για να την αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε ενότητα, βούληση και να περάσουμε στην πράξη. Σήμερα να περάσουμε στην πράξη. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, σήμερα. Και να δράσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ελέγξουμε όπως όλες οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου και να ελέγχουμε τα σύνορά μας αποτελεσματικά. Δεύτερον, η εκπαίδευση εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική για τέτοια θέματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί η τρομοκρατία βρίσκεται στις πόρτες μας. Πρέπει να έχουμε στρατηγική και για την εξωτερική μας πολιτική, προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις στις συγκρούσεις όπως εκείνη τη Συρίας ή της Λιβύης. Εν κατακλείδη, αν όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε με 28, τόσο το καλύτερο. Αν όμως δεν μπορούμε όλοι μαζί, τότε ας αποφασίσουμε μερικοί από μας να δράσουμε. Κάποιες χώρες να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να προχωρήσουν. Η Γαλλία και η Γερμανία, για παράδειγμα, θα πρέπει να βρουν και πάλι την έμπνευση και το όραμα, το οποίο τόσο πολύ λείπουν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. για 1,5 λεπτό η κυρία Ευχαριστώ. στο Πακιστάν χρησιμοποιούνται εξοπλισμένα μη επανδρομένα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα. Βάλουν κατά πολιτών. Ε, συνομίλησαν κάποιοι με παιδιά σε ένα χωριό στο Πακιστάν που είπαν ότι χαιρόμαστε πολύ όταν έχει βαριά συννεφιά και έτσι δεν μπορούν να πετάνε αυτά τα drones και έτσι είμαστε ασφαλείς να παίζουμε έξω. Πρέπει να θυμούμαστε λοιπόν ότι όταν γίνεται ακραία προσπάθεια κατά πολέμης τρομοκρατίας, τα μέτρα δεν στρέφονται κατά της τρομοκρατίας, αλλά σπέρνουν τον τρόμο στους αμαχούς. Τους απλούς αυτούς ανθρώπους, τα παιδιά. Και δεν θα προχωρήσουμε ούτε σπίθαμοι ούτε σπιθαμή στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, να προσπαθήσουμε τη φωτιά να τη σβήσουμε με φωτιά. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να στεγνώσουν πια όλες οι μορφές εξασφάλισης πόρων και όχι μόνο οικονομικών της τρομοκρατίας. Πρέπει να κοιτάξουμε και την Σαουδική Αραβία, την μεταφορά όπλων από εκεί, την ε, τρομοκρατία, την, ε, ε, τους βομβαρδισμούς στους οποίους έχει καταλήξει η Τουρκία εις βάρος του ΠΚΚ αντί να, να βομβαρδίζει το ΝΤΑΕΣ, το Ισλαμικό λεγόμενο κράτος, πρέπει να μην αφήνουμε να χάνονται οι πολίτες γιατί κανείς δεν τους υποστηρίζει. Χρειαζόμαστε στρατηγικές λύσεις, στρατηγικές συμφιλίωσης. Και τελευταία φράση αποδυναμώνονται από αυτές τις ακραίες ε, κατασταλτικές δράσεις οι πολίτες μας. Κυρία Τζέιμς έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ας μιλήσουμε περίφραστα για την κατάσταση. Η τρομοκρατική απειλή είναι στην πραγματικότητα εμφύλιος πόλεμος. Προσπαθεί να διασπείρει το φόβο να φέρει την καταστροφή στις κοινωνίες μας. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ελέγχουν εδάφη οι τρομοκράτες από τα οποία μπορούν να εξάγουν τη βίαιη ιδεολογία τους και έχουν σε τους εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στον Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα, η καλύτερη δυνατότητα που τους προσφέρεται, τους προσφέρεται χάρη στο Σέγγεν για την διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και ακραίας τρομοκρατικής ιδεολογίας όπως και ανθρώπινου δυναμικού. Διευκολύνουν οι κανόνες του Σέγγεν την διακίνηση της χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε δεν πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, να σταματήσουμε τη λειτουργία του Σέγγεν και να διακόψουμε έτσι και τη χρηματοδότηση αυτών των τρομοκρατών. Ε, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Πόλτσακ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η απάντησή μας στις δρομοκρατικές ενέργειες θα πρέπει να είναι αποφασιστική αλλά και ισορροπημένη. Πριν προχωρήσουμε στην εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα εάν οι κανόνες τους οποίους ήδη έχουμε για την καταπολέμηση του φαινομένου εφαρμόζονται σωστά και είναι ικανοποιητικοί. Εξαντλούμε τις δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Οι εκθέσεις του Frontex σαν παράδειγμα δεν πρέπει να αγνοούνται για την είσοδο των μεταναστών. και δεν θα πρέπει εμείς να αφήνουμε να μπαίνουν στην Ευρώπη οι εχθροί της χριστιανικής και ιουδαϊκής μας ιστορίας. Απειλούν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούμεθα να την υπερασπιστούμε. Και δεν θα πρέπει για κοντόφθαλμες πολιτικές ε, για κοντόφθαλμα πολιτικά ωφέλη να αφήνουμε εμείς ε, αυτούς οι οποίοι ελεύθερους, αυτούς οι οποίοι κηρύσουν το μίσος και την ανελευθερία. Θέλουν να καταστρέψουν τις αξίες μας, θέλουν να καταστρέψουν την ιστορία μας. βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη οι οποίες τηρούν μια περίεργη στάση γιατί μεταξύ των άλλων δέχονται και διάφορες μορφές χρηματοδότησης από την Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα. Το ίδιο κάνει και το Αμερικανικό Κογκρέσο. οι Ρώσοι δεν θεωρούν ότι η Τσετσένοι και το Ίσις είναι ο βασικός τους εχθρός, αλλά η Δυτική Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία, χώρες μέλη δεν μπορούν να δράσουν μόνοι τους. Πρέπει να συντονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εθνικές πολιτικές, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία, οι σοσιαλιστές ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, ε, δικαστικές αρχές, τις χώρες μέλη. Ε, με το νέο κέντρο της Europol μπορούμε να έχουμε έτσι ένα ευρωπαϊκό κέντρο, πραγματικά ευρωπαϊκό. Έπειτα πρέπει να καταπολεμηθεί και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, να εναρμονιστούν οι τρόποι ε, συλλογής ε, δεδομένων, και να παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία των τρομοκρατών. Είναι κάτι που να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και όσον αφορά τώρα τη στρατολόγηση από το Ισλαμικό κράτο των μαχητών, πρέπει να αντιμετωπιστεί η ρίζα τη τρομοκρατίας με μια συστημική πολιτική πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση. Η Ευρώπη και οι χωρέ μέλη πρέπει να έχουν περισσότερα μέσα στη διάθεσή του για να χρηματοδοτούν προληπτικά μέτρα σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο σχολείο, στι γειτονιέ, στι επιχειρήσει, αλλά και στο διαδίκτυο. Έχουμε την υποχρέωση με τις δικές μας πολιτικές να δείξουμε ότι οι νέοι μας, όλοι οι νέοι έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τις κοινέ αξίες μας σεβασμού και αλληλεγγύης με όλες τις θρησκείες και με τη μουσουλμανική θρησκεία που είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας κοινότητας. Ευχαριστώ το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κασνοντέψκι. Σας παρακαλώ να σηκώνετε την κάρτα την μπλε λίγο πριν τελειώσει ο προηγούμενος ομιλητής. Οι συνεργάτες μου δεν είναι υπεράνθρωποι. Ο κύριος Κρασνοντέψκι. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέρφους που λένε ότι η τρομοκρατία είναι και ενδοευρωπαϊκή απειλή. Το ξέρουμε ότι ένας στους δέκα στον Ανωμένο Βασίλειο, ένας στους έξι στην Γαλλία πιστεύουν αυτό. Οι χώρες που στέλνουν πολλούς μαχητές πέρα από την Αλβανία και το Σπακιστάν είναι το Βέλγιο, για παράδειγμα όπου βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ή από τη Γαλλία πάνε πολλοί μαχητές ή από την Ελβετία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κύριος ο στόχος για τη στρατολόγηση αυτή είναι νέοι. Νέοι άνθρωποι, παιδιά μεταναστών δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Συχνά είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να ριζώσουν στη νέα κοινωνία στην οποία πήγαν. γυναίκες, παιδιά, οικογένειες που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις ηθικές μας αξίες και πολύ εύκολα καταλήγουν στον θρησκευτικό φανταματισμό. Από την κυρία Βότσμαν, μπλε κάρτα, δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε συνάδελφοι, αναφερθήκατε στο Βέλγιο, τη δικιά μου τη χώρα, ότι εκείνη στέλνει μαχητές, ξένους μαχητές. Εντάξει. Αλλά ευχαρίστως θα ήθελα να ακούσω και από εσά τι θα κάνατε εσείς προκειμένου να λύσετε αυτό το πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ποια δράση θα αναλαμβάνετε εσείς ώστε οι νέοι που μεγαλώνουν στην Ευρώπη πράγματι να μην πηγαίνουν να γίνονται τέτοιοι μαχητές για το ISIS. Κύριε έχετε 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για την απάντηση. Κοιτάξτε, ναι, έχω μια πρόταση για όλους σας. Πολύ συχνά περνάμε ώρες και ώρες με δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα υπάρχουν γειτονιές πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξάλλου, όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι και συνομωτούν για να ετοιμάσουν μια επίθεση. Μήπως κάποια μέρα να πάμε εκεί όλοι εμείς για να δούμε την πραγματικότητα επιτόπου. Και τότε θα μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί ο έλεγχος της πραγματικότητας αποτελεί τη βάση για μια σωστή διάγνωση και στη συνέχεια για την εξέβρεση της σωστής λύσης η πρότασή σας κύριε Κραμψοντέφνη προκάλεσε μια νέα παρέμβαση από την κυρία Βάτμαν. Κυρία Βάτμαν, τι ακριβώς θέλετε. Ευχαριστώ να προσκαλέσω το συνάδελφο μαζί μου να πάμε. Στο Μέχελεν έχουμε φιλελεύθερο ε, δήμαρχο, κανένας δεν έχει φύγει από το Μέχελο. Να δείτε τι τι κάνουμε για την ένταξη των ξένων και για το πώς φροντίζουμε. Οπότε ευχαρίστω να προσκαλέσω τον την επόμενη εβδομάδα. Ελάτε μαζί μου να πάμε στην πόλη του Μάχελεν όπου έχουμε αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Και για τους συναδέρφους που θέλουν επίσης να συμμετάσχουν, ευπρόσδεκτοι. Όλοι θα τα κανονίσετε μαζί, πιστεύω, εξερχόμενοι της αιθούσης. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Γκόμας. ameaça. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες από την τρομοκρατική απειλή. Δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε από την επόμενη επίθεση. Πρέπει με κοινή δράση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη μόνα τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Έχουμε συνεργαστεί σε τομείς αντιμετώπισης προβλημάτων όπως ε, θυμάστε το Ιράκ ε, Ξέρουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν παράλληλα φαινόμενα όπως το λαθρεμπόριο όπλων και το λαθρεμπόριο καυσίμων και υπάρχει και ρόλος αμφισβητήσιμος από πλευράς ορισμένων χωρών όπως η Τουρκία και το Κατάρ. Θα πρέπει να βρούμε επίσης τρόπους αποτελεσματικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες έτσι ώστε να δημιουργηθούν ε, συγκεκριμένες περιοχές ελεύθερες και ελεγχόμενες με το τέλος του Σέγγεν και με νέους τείχους δεν πρόκειται να θέσουμε τέρμα στην, βαβαρία, στην βαρβαρότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο συλλέγοντας τις σωστές πληροφορίες. Ε, δεν έχουμε όμως πολλές φορές την δύναμη να αντιπαρατεθούμε με τους προπαγανδιστές ε, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απορριζοσπαστικοποιήσουμε τους νέους Ευρωπαίους οι οποίοι υποκύπτουν στα κηρύγματα του μίσους. Νομίζω ότι αν δεν είμαστε ενωμένοι το μόνο που θα κάνουμε είναι να βοηθάμε τους τρομοκράτες και να λειτουργούμε εις βάρος των δυστυχισμένων αυτών που προσπαθούν να ξεφύγουν από εκεί. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο κράτος δικαίου, στους κανόνες της δημοκρατίας, θα πρέπει να υπάρξουν σωστές εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές στον τομέα της ασφάλειας. Πρέπει να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Μας έχετε μια μπλε κάρτα από την κυρία Ουφσκοκ. Τη δέχεστε? You have a blue card. Παρακαλώ κυρία Ουφσκοκ, έχετε 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Eh, eh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γκόμες τι έχει να πει στη σχέση με τα όσα συζητήθηκαν νωρίτερα και με τον κύριο Κρασνοτεύσκη στη Σουηδία. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνδρες που έφυγαν για να πολεμήσουν στις τάξεις του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους. Υπάρχουν πολλοί νέοι, άνδρες και γυναίκες, που φεύγουν από τις χώρες τους και φαντάζομαι ότι θα ήταν λιγότερες αυτές τις δραστηριότητες αν δεν είχαν ανάγκη να φύγουν. Well, my country στα αγγλικά. Η χώρα μου έχει πει ότι θα υποδεχθεί έως και 5.000 τους προσεχείς μήνες πρόσφυγες, οι οποίοι όμως δεν έρχονται γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα. Όσοι έφτασαν όμως στην Πορτογαλία, την χάνουν πλήρους υποστήριξης και δυνατοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η πρόσβαση στην εργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, πέραν άλλων ζητημάτων. Ο η κοινωνική ενσωμάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ό,τι πολιτικές έχουν υιοθετηθεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδηγούσαν στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Και ιδιαίτερα αυτό συνέβη σε σχέση με τις κοινωνίες και τις κοινότητες των μεταναστών. Αυτό έσπρωξε τα παιδιά μας στα σύνορα να πάνε να πολεμήσουν εναντίον μας. Παράκληση και η ερώτηση και η απάντηση να μην υπερβαίνουν τα 30 δεύτερα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Γερμανία μόνο οι τρομοκρατικές ε, πράξεις έχουν τριπλασιαστεί. Ε, γίνονται πολλές ε, δίκες εις βάρος των μαχητών του Ισλαμικού λεγόμενου που έχουν δικτυωθεί. Στις 7 Ιανουαρίου, την επέτειο του Σαρλί Επτό συγκεκριμένα, δολοφονήθηκε στο Παρίσι ένας, ε, μάλλον πυροβολήθηκε στο Παρίσι από, την, από τους αστυνομικούς ε, ένας που ονομάζεται Μπέλγατσέμ, ο οποίος τους επιτέθηκε με ε, πέλεκη, ο οποίος διέμενε στη Γερμανία με επτά διαφορετικές ταυτότητες, είτε γεωργιανός, είτε τινήσιος, είτε σύρος, είχε διαφορετικές ταυτότητες. Έζησε λοιπόν στη Γερμανία και, και φαίνεται ότι εκεί είχε διαπράξει μια σειρά από αδικήματα, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την κατάχρηση κοινωνικής πρόνοιας, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ε, ε, κλοπές κτλ. Ήταν το ε, διαμέρισμά του γεμάτο με σύμβολα του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους. Παρόλα αυτά, αυτός ο Μπελγκατσέμ μπόρεσε να κινηθεί ελεύθερα από τη Γερμανία στη Γαλλία, παρότι είχε και το μητρό αυτό. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. 1,5 λεπτό ο κύριος Βάιντε Χόλτσερ. Grundsätzlich. Κατά βάση, οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, απειλητικές, αποτρόπες, με στόχο να αποσυντονίσουν, να αποθεμελιώσουν τις κοινωνίες μας. Ο αγώνας κατά αυτών των τρομοκρατικών απειλών είναι απαραίτητος, είναι σημαντικός, αξίζει όλη μα την προσοχή. Οι τρομοκρατικέ αυτές απειλέ, η τρομοκρατική αυτή απειλή έχει όμως όνομα. Ντάεσ, ISIS, Ίκυλ, αυτό πρέπει να συζητούμε. Δεν μπορούμε τη συζήτηση να την ε, εκμεταλλευόμαστε για πολιτικές αντιπαραθέσεις ε, λαϊκού, λαϊκιστικού τύπου. Εδώ λαμβάνονται μέτρα που έχουμε συζητήσει και στο Κοινοβούλιο όπως η έκθεση για την απορριζοσπαστικοποίηση ή άλλη για το PNR, την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους επιβάτες πτήσεων, αν και δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμη όλο και μεγαλύτερη συσσόρευση προσωπικών δεδομένων, εν πάση περιπτώσει όμως έχει γίνει η συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να μπορούμε να αναλάβουμε δράση βράχη πρόθεσμα. Πρέπει να αναλογιστούμε εάν τα δεδομένα αυτά την χάνουν σωστή ανάλυση ή συλλέγονται με το σωστό τρόπο. Ε, πρέπει να έχουμε πιο κατάλληλα καταρτισμένο και με καλύτερο ε, υποστήριξη προσωπικό στις αστυνομικές μας αρχές. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών ε, συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών των κρατών μελών. Ίσως δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, αλλά κύριε Επίτροπε πρέπει να κοιτάξουμε να ε, τους πείσουμε να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. για ένα λεπτό Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2015 ήταν η χρονιά με τα περισσότερα θύματα από την τρομοκρατία, μετά βέβαια από το 2004 στη Μαδρίτη. Θα την ξαναπάθουμε, αν δεν φροντίσουμε. Πού και πότε δεν ξέρουμε βέβαια. Έχουμε κράτος δικαίου και ελευθερίες στην Ευρώπη, που δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο βωμό κάποιας ασυντόνιστης εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό και πρέπει με ψυχραιμία και με σοφία να προχωρήσουμε και να μην κάνουμε το σφάλμα να νομίζουμε ότι οι ξένοι, οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφαλειά μας. Ούτε με πανικό και με φόβο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να συμπληρώσουμε το Σέγγεν με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή για την φύλαξη των εξωτερικών ε, συνόρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων. Αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Να συμπληρωθεί το ποινικό ευρωπαϊκό δίκαιο με μια ευρωπαϊκή υπηρεσία αστυνομία και με την προστασία των θυμάτων. Και τέλο, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρέπει. Διερμηνία. Ποια διερμηνία ακριβώ. Δεν έχετε διερμηνία. Πρόβλημα. Θα σας δώσω το χρόνο. Συνεχίστε την ομιλία. Έχετε ακόμη μισό λεπτό. Μπορείτε να συνεχίσετε. May I proceed now? Yeah, yeah. You can proceed. El camino, Έλεγα λοιπόν ότι ο σωστός δρόμος είναι να ξέρουμε ότι οι τζιχαντιστές και ο κοινωνικός ε, αποκλισμός συνδέονται. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τον αποκλεισμό και τις ανισότητες. Πρέπει να μιλήσουμε με τις κοινότητες οι οποίες επίσης έχουν πληγεί από την καταστολή που ακολούθησε. Δεν πρέπει να υπάρχουν τόσε ανισότητε στην Ευρώπη. Να μην υπάρχει αποκλεισμό, κάτι το οποίο οδήγησε σε πάρα πολλού οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ευρώπη αλλά και σε Ευρωπαίου αυτόχθονε να γίνουν τρομοκράτε. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλάρ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Μαμίκιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως έχουν ε, ανέβει πολλές εθνικιστικές ομάδες και χωρίζουν τους Ευρωπαίους μεταξύ τους. Η τρομοκρατία δεν έχει σύνορα όμως, είναι και τοπική αλλά γίνεται και όλο πιο ριζοσπαστική από ό,τι κατά το παρελθόν. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρηνική λύση. Ο μόνος λογικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη και να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα είναι να αλλάξουν οι πολιτικές μας όσον αφορά την ένταξη, να εμποδιστούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, των τρομοκρατών. Και βέβαια χρειάστηκε μια πιο επιθετική πολιτική από τη δικιά μας την πλευρά για εκείνους οι οποίοι ανοιχτά μέσω της θρησκείας προχωρούν στην προπαγάνδα, είτε πρόκειται για τη Σοδική Αραβία είτε Δεν προτείνω εδώ να καταργήσουμε τις βασικές μας αξίες. Αλλά λέω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών, να μην τους βάζουμε σε κίνδυνο πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω δεχθεί έξι αιτήματα. Επειδή η συζήτηση έχει ενδιαφέρον, τα κάνω δεκτά όλα. Προχωρούμε με τον κύριο Μπόγκοβιτς. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ε, τους λόγους για τους οποίους ε, ε, υπάρχει το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Καταρχάς πάρα πολλοί νέοι από την Ευρώπη είναι απογοητευμένοι γιατί δεν έχουν μέλλον. Ζούνε σε γκέτο κάτω από πολύ καλές συνθήκες και εκεί ακριβώς η τρομοκρατία φυσικά έχει πολλά να κερδίσει. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το Αφγανιστάν, η Συρία, η Λιβύη έχασαν τις δικτατορίες εισαγωγικά τις οποίες είχαν και αυτό συνολικά αποσταθεροποίησε ε, την περιοχή γενικότερα. Ταυτόχρονα έχουμε και το φαινόμενο χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ενεργειών από πολλές αραβικές χώρες. Και αυτό έχει συνέπειες και για την Ευρώπη. Εδώ έρχεται το θέμα της καλύτερης και πληρέστερης ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Πρέπει να φανούμε ευφυείς και αποτελεσματικοί και δεν θα πρέπει εμείς να επιτιθέμεθα σε τίμιους Ευρωπαίους, σε ειλικρινείς τίμιους πολίτες, το οποίο κάνουμε φοβάμαι μέσω της νέας οδηγίας για τα μικρά όπλα λήξη της ομιλίας δεν το δέχομαι. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να καταλαβαίνουν τι λέει ο μιλητής πριν τελειώσει. Παρακαλώ το αίτημα για μπλε κάρτα να διατυπώνεται έγκαιρα, αλλιώς δεν θα το κάνω δεκτό, πολύ περισσότερο που είμαστε στη διαδικασία του ΚΑΤΖΙΑΙ. Παρακαλώ, το λόγο έχει η κυρία Γκραπίνη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, σε περίοδο κρίσης φαίνεται αν μια οικογένεια, μια ένωση, μια κοινωνία μπορεί να αντισταθεί. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών μας. Πρέπει αυτή να είναι προτεραιότητα του Συμβουλίου όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπουργός των Κατοχωρών μας είπε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το μίσος κατά των μουσουλμάνων. Ναι, αλλά πρέπει και να προτείνετε και να προβάλλεται λύσεις ώστε οι μουσουλμάνοι να αποδέχονται τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, να αποδεχθούν τον τρόπο ζωής μας, εάν χρειάστηκε να έρθουν μέχρι εδώ λόγω των δυσκολιών ή των συγκρούσεων. Εδώ είναι το σφάλμα όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση με τους ε, πρόσφυγες πρέπει να γίνει περισσότερη ε, προσπάθεια επικοινωνιακή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή όπως και το Συμβούλιο πρέπει να προσφέρουν ένα σαφές σχέδιο για τη διαχείριση του προσφυγικού και των οικονομική του της οικονομικής μετανάστευσης για τους πολίτες. Δεν μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει με το δικό του τρόπο την ε, προσφυγική κρίση, ούτε να φτάσουν βέβαια οι κάτοικοι ολόκληρων κρατών να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα συνεκτικό κείμενο ε, γιατί μπορεί μια πλειοψηφία που δεν, διαχειρι... δεν τη χάνει σωστής διαχείριση να ανατρέψει ολόκληρες κοινωνίες. Ε, η καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής θα γίνει αποτελεσματική μονάχα όταν αναγνωριστεί η αφετηρία της, που είναι η προσχώρηση μεγάλων μερίδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων της Μέσης Ανατολής στον φονταμενταλισμό. Ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια αυτού του πολιτικού και κοινωνικού φαινομένου επιπλέον πρέπει να αναγνωριστεί ο τυχοδιοκτισμός με τον οποίο κάποια ευρωπαϊκά κράτη και πρωτίστως η γαλλία παρεμβαίνουν στρατιωτικά στη μέση ανατολή από το. 2011. χιλιάδες τέλος οι ίδιες οι χώρες της ευρώπης οφείλουν να αναγνωρίσουν την τεράστια αποτυχία των πολιτικών ένταξης των μουσουλμάνων να επανακινήσουν τα σχετικά προγράμματα που εγκαταλείφθηκαν για ιδεολειπτικούς λόγους μετά τη δεκαετία του 1980 και να απεμπολίσουν τις ρητορικές μίσους από την πολιτική αντιπαράθεση που αυτοεκπληρώνουν τη θεωρία της πολιτιστικής και πολιτισμικής σύγκρουσης. ήρθε η ώρα η ευρώπη να ακολουθήσει ένα άλλο υπόδειγμα στις διεθνείς και διαπολιτιστικές σχέσεις με τα κράτη της μέσης ανατολής και της βορείου αφρικής. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μαρίνιο Επίντου. Κύριε Φαρία, θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα πάρετε και εσείς. Θα μιλήσετε και οι δύο. Μην ανησυχείτε. Είπα ότι θα μιλήσετε όλοι. I repeat it. O combate ao terrorismo. That you will speak all together. After, after two speakers. Παρακαλώ κύριε Μαρίνιο Επίντου έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ξεκινάει από τη μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φανετισμού. Και συνεχίζεται με τον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και υπέρ των ατομικών ελευθεριών. Κυρίως για την ελευθερία μετακίνησης των Ευρωπαίων μέσα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πιστεύει και αγωνίζεται όπως λέει ο Τζορτ Στάινερ, και έδωσε τα φώτα και όλες οι θρησκείες αγωνίζονται υπέρ του πολιτισμού. Από τις τρεις μονοθυστικές θρησκείες φτιάχτηκε η Ευρώπη. Δεσμό, χριστιανισμό και Ισλάμ. Προσπαθούμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Τώρα όμως, με άλοθη την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα βάζουμε με μια θρησκεία. Ε, πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, η καταπολέμηση της ριζασφαστικοποίησης πρέπει να είναι και ο αγώνας κατά της μυσαλλοδοξίας που δυστυχώς ανεβαίνει στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα αίτημα για μπλε κάρτα από τον κύριο Τσαμπάσκι, όπως όμως με ενημερώνει συνεργάζομαι ο κύριος Τσαμπάσκι έχει ήδη μιλήσει για το θέμα. Αυτό... Κύριε Τσαμπάτσκι, καθίστε κάτω, βάλτε τα ακουστικό σας να ακούσετε τι θα πω. Please sit down and put your uh, translation in your ear. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχετε μετάσχει στη συζήτηση και επειδή είμαστε στη διαδικασία του catch the eye, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να σας δώσω το λόγο με το δικαίωμα της μπλε κάρτας. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε τη δυνατότητα ομιλητών που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο να μιλήσουν και αυτοί. Σας παρακαλώ λοιπόν να το καταλάβετε και να μην επιμείνετε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Τόματσιτς για ένα λεπτό. Hvala lijepa. 2015. su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta, a prema posljednjim informacijama Δυστυχώς οι τρομοκράτες εξακολουθούν να εμπλουτίζουν τις ε, δυνάμεις τους και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε με πανικό. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας αυξάνοντας τα μέτρα ασφαλείας και προσπαθώντας να προλάβουμε αυτούς οι οποίοι συνομωτούν εναντίον της δημοκρατίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δράσουν πιο αποτελεσματικά και να μην περιμένουν από υπερεθνικές μορφές συνεργασίας της λύσης. Η ασφάλεια των πολιτών μας είναι ο απόλυτος στόχος ο ανώτερος στόχος. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από αυτό. Και Φαρία, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ε, Τουρκία και την Πουρκίνα Φάσο όχι μόνο ενισχύουν την ε, τρομοκρατική απειλή, αλλά καταδεικνύουν και τον υπερεθνικό της χαρακτήρα, την ανάγκη να δοθεί μια συντονισμένη απάντηση. Στον αγώνα λοιπόν κατά της τρομοκρατίας πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει όχι μόνο τη συνεργασία της στρατιωτικά θέματα στα θέματα ασφάλισης, αλλά και να καταπολεμήσει τη ριζοσπαστικοποίηση, να καταπολεμήσει την χρηματοδότηση, τα επιμελητιακά μέσα που έχουν οι μαχητές στη διάθεσή τους, για να καταπολεμήσουν τον τρόπο ζωής μας, για να μας αφαιρέσουν τις ζωές μας. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τους Πεσμέργα, παραδείγματι, μαχητές, οι οποίοι όταν έρχονται στην Ευρώπη, αν τραυματιστούν και έρθουν στην Ευρώπη να ε, θεραπευτούν σε θεραπευτήρια, ε, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν πολύ ακριβά νοσήλια. Πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους άμαχους, μάλιστα κύριε Πρόεδρε, να μετατραπούν σε παρεπίπτωτα θύματα της τρομοκρατίας. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου και η διαδικασία του Eye, Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Έλεγα να αποφασιστώ τις ευκαιρίες για να θυμηθώ λίγο τα ελληνικά μου, το γεγονός ότι προεδρεύεται, αλλά προτιμώ να μιλήσω στα ε, αγγλικά και ευχαριστώ για αυτό. Ε, ε, Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, παρακολούθησα την συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Κανένας δεν μένει αδιάφορος απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα και πιστεύω ότι σε αυτήν εδώ την Ολομέλεια προσπαθούμε να ενισχύσουμε την συνειδητοποίηση, την διαδικασία συνειδητοποίησης του προβλήματος και την ανάγκη που υπάρχει για να το καταπολεμήσουμε. Για την κυρία Σαρτζεντίνη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ερώτησή σας, αν και τα διευκρίνησα κάπως στην αρχή της ομιλίας μου. Οι τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμα και αυτές που δεν οργανώνονται ή δεν προέρχονται από ένα ευρύτερο δίκτυο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο κοστίζει χρήματα για την προετοιμασία, για τα όπλα, για τα ψευδή έγγραφα, τα παραποιημένα έγγραφα, Νομίζω ότι ε, το κόστος ε, είναι πολύ υψηλό και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποδείξω εγώ την προσπάθεια την οποία κάνουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την επιθυμία μας να διασφαλίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχουν υπάρξει βήματα προόδου έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση στα θέματα ασφάλειας. Όμως δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας γιατί η τρομοκρατική απειλή είναι πάντα παρούσα. Η απειλή είναι απτή και απαιτούνται δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα αλλάξουν την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε ημέν τις προσπάθειες των δε για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα ευρωπαϊκά όργανα, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές αρχές, οι δυνάμεις επιβολής τάξης, οι δυνάμεις συλλογής πληροφοριών, όπως επίσης και οι δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα επανέλθω σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Τα κράτη-μέλη είναι ανάγκη να εμπιστεύονται το ένα το άλλο περισσότερο. Είναι ανάγκη να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες. Όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις ευρωπαϊκές επιρροσίες. Προσωπικά πρέπει να πω εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο της συνεργασίας μέχρι τώρα δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω, κρατούν τις περισσότερες και καλύτερες από τις πληροφορίες που συλλέγουν για τον εαυτό τους. Έχει φτάσει η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα ακόμη. Η προσπάθειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει και θα διπλασιάσει τις προσπάθειές της ε, το 2016 θα υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις από πλευράς της Επιτροπής, ιδιαίτερα όπως είπα στο θέμα της χρηματοδότησης. Υπολογίζω στη δική σας στήριξη. Απαιτείται να προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Απαιτείται να προωθήσουμε ευρωπαϊκές λύσεις γιατί έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, την τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υποστήριξή σας. Το λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου ο κύριος Κούντερς. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για την τρομοκρατία. Θα αρχίσω λέγοντας ότι η τρομοκρατία είναι ένα τέρας με πολλά πρόσωπα και απαιτεί πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Δεν φτάνει μία για να καταστρέψουμε την τρομοκρατία. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και την αισθηματική φόρτιση που είχαμε στην σημερινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μην ξεχνάμε τα θύματα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά. Κάτι που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά και για να τους τιμήσουμε σας διαβεβαιώνω ότι και το Συμβούλιο ενεργοποιείται ιδιαίτερα προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, αλλά επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν απλοποιούμε το θέμα της τρομοκρατίας, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο που είναι σαν το χταπόδι, Λερνέα Ήδρα, Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται καταστολή, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Αν δεν συμφωνήσουμε για την πολιτική ατζέντα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άκουσα την πολιτική ελίτ. Κάποιο, ο κ. Μπανάνα, νομίζω, αναφέρθηκε σε αυτό. Εγώ εδώ εκπροσωπώ το Συμβούλιο, όχι την Ολλανδική κυβέρνηση. Το Συμβούλιο. Και στο Συμβούλιο εδρεύουν κυβερνήσει από διαφορετικέ πολιτικέ αποχρώσει. Δεν ξέρω, 100.000 το χρόνο βγάζετε, δεν ξέρω, με κάθε σεβασμό προς τους ευρωβουλευτές και οι υπουργοί πληρώνονται βέβαια, αλλά αν εσείς είσαστε από την πολιτική ελίτ, είμαι και εγώ τότε. Δεν πρέπει λοιπόν κάποιοι εδώ να νιώθουν ότι εκπροσωπούν περισσότερο τον κόσμο από ό,τι άλλοι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικέ απόψει μεταξύ μα, αλλά δεν θα κάνουμε τη συζήτηση απλοποιώντα. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε την απλοποίηση τη τρομοκρατία. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Και αν λοιπόν εμείς αναλύσουμε σωστά το τι συμβαίνει και συνεργαστούμε, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν πρόκειται ο καθένας να θέλει ε, το δικό του το κομματάκι μόνο, μα αυτό ακριβώ ψάχνουν οι τρομοκράτες από εμά. Τότε θα χάσουμε. Τι είναι τρομοκρατία? Μια στρατηγική που εμφυσά το φόβο στους πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ας μείνουμε ψύχρεμοι. Ας δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, και πρόληψη και καταστολή και συνεργασία και ε, καταπολέμηση ε, του Ισλαμικού κράτους. Πολύ σωστά είναι όλα αυτά. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το Συμβούλιο. Είχαμε μια διάσκεψη πριν από 10 μέρες στις κάτω χώρες. Είχε να κάνει με το παγκόσμιο συνασπισμό κατά του ISIS. Μα περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να συνδυάσουμε την εμπιστοσύνη με την ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον για να γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας. Και γιατί δεν συμβαίνει αυτό πάντα και γιατί θα έπρεπε να συμβαίνει παραπάνω το πατόλι εδώ και το Συμβούλιο συμφωνεί. Είναι όμως κατανοητό το τι σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών και το πήραμε αυτό το μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεργασία των υπηρεσιών συμμόρφωση του νόμου, ε, μυστικέ υπηρεσίες, κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και να ενισχύσουμε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας. Η καλύτερη απάντηση από τι κοινωνίε μα είναι η αντοχή και η στήριξη των αξιών μας υπέρ του κράτους δικαίου και των ελευθεριών. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Και μετά περνάμε σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ναι, το θέμα είναι η εφαρμογή βέβαια των ρυθμίσεων που εγκρίνονται. Το Συμβούλιο δουλεύει σε διαφορετικέ συνθέσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μας. Πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία με... φτάσαμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο δηλαδή, όσον αφορά την οδηγία για το Ευρωπαϊκό PNR. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό PNR θα μπορέσει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας πραγματικά. Πρέπει να υλοποιηθεί. Και έχουν εγκριθεί μέτρα επίσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και για το πώς τα στοιχεία από το PNR θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών όταν χρειάζεται πίσω. Τώρα, το θέμα της χρηματοδότησης, του λαθρεμπορίου όπλων, η καταβλησμή με τα κέντρα εκπαίδευσης ε, τρομοκρατών στο εξωτερικό, αυτά είναι επίσης πράγματα τα οποία πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε και να παρακολουθούμε τους υπόπτους για οργανωμένο έγκλημα. Αναφερθήκατε στη Συμφωνία PNR και στην Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων, τη σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Ναι, το ξέρω και εγώ, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Το έχουμε υπόψη μας. Έχουμε απαντήσει ότι αυτή η σχέση πρέπει να καλυφθεί από μια νέα ρύθμιση, η οποία θα εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και το Συμβούλιο έχει ήδη προχωρήσει και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ό,τι δράση χρειάζεται ώστε να εγκριθούν τα απαραίτητα μέτρα όσο γίνεται πιο γρήγορα και το γλωσσικό ζήτημα πρέπει επίσης να καλυφθεί ώστε το κείμενο να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο και σωστό. Τα θεσμικά μας όργανα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Έχετε τη δέσμευσή μου επ' αυτού για να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έχουμε φτάσει σε συμφωνία και για το PNR και για την προστασία δεδομένων. Δεν θα καθυστερήσουμε παραπάνω. Συνεργασία χρειάζεται, υποχρεωτική ή όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι βάση του 4.2 της συνθήκης η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα της κάθε χώρας μέλους. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει και μια συνεργασία και εμπιστοσύνη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομική βάση γι' αυτό για τις ανησυχίες σας, για την ισορροπία μεταξύ των δύο. Εντάξει, είναι εύκολο να είμαστε στην καταστολή για την προστασία του ιδιωτικού βίου να πούμε ότι θέλουμε μια ισορροπία. Ναι, το Κοράνι δεν έχει καμιά σχέση με τους φανταματελιστές και το Ισλάμ. Εντάξει, δεν, τα λόγια δεν βοηθούν. Το Συμβούλιο δουλεύει για συνδυασμένε προσπάθειες όσον αφορά την πρόληψη, αλλά πρόληψη και καταστολή. Το κράτος δικαίου φυσικά και θέλουμε να το τηρούμε και να προστατεύουμε τις αξίες μας. Ό,τι μέτρα παίρνουμε πρέπει να γράφονται πάντα στα πλαίσια των όσων προβλέπουν οι αξίες μας και το κράτος δικαίου. Αυτό όμως, ναι, σημαίνει πρόληψη. Πρόληψη δεν είναι μια ήπια πολιτική. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και έχει να κάνει και με τις οικονομικές δυνατότητες και τις διακρίσεις δεν πρόκειται μόνο για την άμυνα. Πρέπει να παρακολουθούμε ολόκληρη την αλυσίδα ριζοσπαστικοποίησης. Το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι η απάντηση. Πολλοί είπαν εδώ πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και συγχρόνως λέτε χρειαζόμαστε περισσότερη διεθνή συνεργασία. Ε, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαν στη συνάντησή μας και άλλες χώρες που το γνωρίζουν και γι' αυτό και χρειάζεται συνεργασία και με τρίτες χώρε στη Βόρεια Αφρική και αλλού. Το χρονοδιάγραμμα για τη δικιά μας συνεργασία τώρα, και καλό είναι που έχουμε τέτοιες συζητήσεις συχνά μαζί, ως εκτελεστικό σκέλος πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εσάς έχουμε έναν εχθρό ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερα και αυτό δεν έχει να κάνει με τα σύνορα. Γι' αυτό χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ό,τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ μας δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση της αποτελεσματικότητά μας για την καταπολέμηση της απειλής αυτής. Ευχαριστώ. Η συζήτηση Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στην προφορική ερώτηση της Επιτροπής με θέμα την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Εμπορικών Σχέσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κύριος Λάγκε, συντάκτης της ερώτησης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε,